Άλλη ανακοίνωση. Ο πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες την Σοσιαλιστική και Δημοκρατική και το ΙΣΙΑΡ ορισμένα αιτήματα για διορισμούς σε επιτροπές και σε μια αντιπροσωπεία. Αυτές, αυτοί οι διορισμοί θα περιλαμβάνονται στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης. Εάν δεν ε, υποβληθούν παρατηρήσεις μέχρι την έγκριση των πρακτικών, οι διορισμοί αυτοί θα θεωρηθεί ότι εγκρίνονται.